Καλημέρα σα Θα ξεκινήσουμε τη σημερινή συνεδρίαση. Το πρώτο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Έχετε κάποιες τροποποίησεις ε, στην ημερήσια διάταξη. Νομίζω ότι έχει γίνει μια γενικευμένη συνένεση εδώ για την έκθεση της ε, συναδέλφου Ιώτοβα για, την, ε, για τον έξινο πόντο και επίσης υπάρχει και μία αλλαγή κατόπιν αιτήματος των σοσιαλιστών για μία γραπτή ερώτηση για τα ε, βιωσιμότητα της αλληλείας Εγώ ε, δέχτηκα να συμπεριληφθεί το σχετικό σημείο στην ημερήσια διάταξη, αλλά να σας πω ότι το άρθρο 117 σημείο 3 του κανονισμού στο οποίο βασιστήκαμε για να γίνει αυτό το αίτημα δεν είναι το κατάλληλο σημείο, γιατί το 117 σημείο 3 αναφέρεται απλώς ε, στις ερωτήσεις οι οποίες δεν έχουν λάβει απάντηση από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής και είναι αρμοδιότητα τη Επιτροπή μα. Κανένα από τα δύο λοιπόν αιτήματα δεν πληρούνται εδώ. Δεν θα ήθελα να ε, προχωρήσω άλλο το θέμα γιατί όταν έδωσα την έγκρισή μου δεν είχα εξετάσει το σχετικό άρθρο αλλά σας παρακαλώ μη μου ξαναζητήσετε κάτι το οποίο δεν είναι ορθό γιατί θα αρνηθώ στο μέλλον. Αν δεν υπάρχουν λοιπόν άλλες ενστάσεις ε, μπορούμε να θεωρούμε ότι είναι ε, η εμερήσια διάταξη. Να σας πω ότι ως συνήθως η συνεδρίαση αυτή μεταδίδεται ζωντανά στο διαδίκτυο. Έγκριση των πρακτικών της συνεδρίας 24ης και 25ης Μαΐου του 2011. Εάν στη διάρκεια της συνεδρίασης δεν παρουσιαστούν αντιρρήσεις, θα θεωρήσουμε ότι εγκρίνονται και τα πρακτικά. Δεν έχω καμία ανακοίνωση να σας κάνω στο σημείο 3. Το σημείο υπαριθμών 4 είναι η έκθεση της κυρίας Ιώτοβα για το μέλλον ε, της Αλίας στη Μαύρη Θάλασσα και τη διαχείριση των αλληλευτικών δραστηριοτήτων. Το θέμα το έχουμε συζητήσει. Σήμερα θα κάνουμε μια συζήτηση για τις τροπολογίες που κατατέθησαν καταρχάς και μετά θα ψηφίσουμε απευθείας ε, την έκθεση. Καταρχάς λοιπόν να δώσω το λόγο στην κυρία Ιώτοβα και στη συνέχεια στους ε, συναδέλφους που έχουν καταθέσει τροπολογίες για να μας εξηγήσουν τους λόγους για τους οποίους κατέθεσαν τις τροπολογίες και να δούμε και λίγο τις συμβιβαστικές τροπολογίες ε, οι οποίες ε, εξ όσων γνωρίζω έγιναν αποδεκτές από τις περισσότερες πολιτικές ομάδες. Κυρία Ιώτοβα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε οι τροπολογίες για την έκθεση σχετικά με την τρέχουσα και μελλοντική διαχείριση της αλίας των εύξηνων πόντων έχουν ήδη κατατεθεί. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους αυτούς που κατέθεσαν τροπολογίες και βεβαίως και κατά τις συζητήσεις που έγιναν στο παρελθόν βεβαίως έχουμε ακούσει τις απόψεις όλων ε, ακούσαμε τις θέσεις των εμπειρογνωμόνων από τη Βουλγαρία αλλά μιλήσαμε και με τους εκπροσώπους της ε, Τουρκίας και άλλων χωρών στο στο και τον γειτονικών χωρών της ε, Μαύρης θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κύριο Ιωάννη Τσουκαλά για τις ε, τροπολογίες που κατέθεσε και τον κύριο τον Σκιώδη, εισηγητή δηλαδή. Οι τροπολογίες ειδικά του κυρίου Τσουκαλά αναφέρονται στις συζητήσεις, στη σημασία των συζητήσεων με τις χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες ενέχονται στην όλη υπόθεση λέγεται ότι η κοινή αρχή πρέπει να είναι πιο ενεργή, ότι πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα και ότι θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν όλα τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας για να ενισχύσουμε τη σχέση μας με την, ε, τις άλλες χώρες του εύξηνου πόντου. Συμφωνώ απόλυτα με τον ε, σκιώδη συγητή για τα θέματα αυτά, για αυτά που αναφέρει στις τροπολογίες του. Βεβαίως δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και την ιδέα ιδέα της ειδική αρχής για τον εύξηνο πόντο. Πρέπει να αποδώσουμε σίγουρα μεγάλη σημασία γενικότερα στη Μαύρη Θάλασσα ε, και ειδικότερα στην αρχή αυτή. Οι χειμερινοί αγώνες της ε, ε, στο Σότσι ξέρουμε ότι έχουν ε, ότι απαιτούν ε, κατασκευές, έργα και τα στην περιοχή. Συμφωνούμε μέχρι εδώ. Αλλά από εκεί και πέρα η οικολογία των περιοχών πώς θα επηρεαστεί από τα έργα και τις κατασκευές αυτές θα ήθελα να επισύρω την προσοχή σας στην ε, τροπολογία του κυρίου Τσουκαλά για την ε, αιτία επίσης της αλίας και της ε, παράνομης εντός εισαγωγικών αλίας. Αυτή είναι πολύ σωστή παρατήρηση. Από την άλλη μεριά έχουμε προβλήματα μεταξύ Βουλγαρίας και Ρουμανίας ε, και περιμένουμε να και την ε, Κομισιόν να ε, κάνει παρατηρήσει σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού 2371. Υπάρχουν πολλά προβλήματα τα οποία πρέπει να επιληθούν και εδώ ο κύριος Κάντεκ προτείνει να φτιάξουμε μια ευρωπαϊκή ε, ακτοφυλακή τρόπον την Εγώ νομίζω ότι δεν είναι κακή ιδέα αυτή. Επίση, συμφωνώ με όλους αυτούς που λένε ότι πρέπει να ενισχύσουμε και την την οικονομία αν θέλει της ευρωπαϊκής αγοράς η οποία ε, ενισχύεται και χρειάζεται και τις εισαγωγές προϊόντων από τρίτες χώρες. Υπάρχει επίσης συμβαστική πρόταση, συμβαστική τροπολογία 5, η οποία, ε, την οποία αξίζει να... προσέξουμε η τροπολογία αυτή είναι πάρα πολύ καλή και θα ήθελα γι' αυτό να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά όλους αυτούς που ζητούν την συνεργασία όλων των επιστημονικών και άλλων αρχών στην περιοχή η οποία συνεργασία μπορεί να μας ε, βοηθήσει να προχωρήσουμε. Ο κύριος Τσουκαλάς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την εισηγήτρια για την αξιόλογη έκθεση που παρουσίασε, καθώς επίσης και για την επικοδομητική συνεργασία και τις συμβαστικές προτάσεις που εισηγήθηκε. Η Μαύρη Θάλασσα αποτελεί αδιαμφισβήτητα μία από τις πιο δυναμικές ημίκλειστες θάλασσες με σημαντικό περιβαλλοντολογικό αντίκτυπο στους πληθυσμούς των χωρών που την περιβάλλουν καθώς βρίσκεται σε σημαντικό γεωστρατηγικό σημείο και εκτείνεται πέραν των ευρωπαϊκών ορίων. Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης περιοχής, είναι σημαντικό ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ξεκινά συζήτηση για τις ανάγκες τόσο της θαλάσσιας βιοποικιλότητας όσο και για τον αλλιευτικό κλάδο της περιοχής. Οι τροπολογίες που κατέθεσα αποσκοπούν στο να καταστήσουν το κείμενο πιο συνεκτικό, ολοκληρωμένο και ρεαλιστικό και οι βασικότερες ιδέες θα μπορούσαν να συνοψιστούν ως εξής. Πρώτον, συμφωνώ με την εισηγήτρια ότι λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας θα πρέπει να λαμβάνεται περισσότερο υπόψη κατά τη συζήτηση για τη χάραξη της ευρωπαϊκής ελληνευτικής πολιτικής. Θεωρώ όμως ότι η δημιουργία ενός χωριστού φορέα τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή δεν θα επιφέρει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα όσον αφορά την προστασία της θαλάσσιας βιοπικιλότητας και την ευημερία των αλλιέων. Δεν είμαι εναντίον της ιδέας μιας νέας οργάνωσης, αλλά η ανάγκη αυτή θα πρέπει να εξεταστεί σε πιο μακροπρόθεσμη βάση. Οι σχετικές συμβιβαστικές που έχουν προταθεί με βρίσκουν απολύτως σύμφωνο. Δεύτερον, όσον αφορά τον ορισμό ειδική γραμμής προϋπολογισμού για τη Μαύρη Θάλασσα, θεωρώ ότι μια παρόμοια πρόταση δεν μπορεί να υποστηριχθεί εν μέσω της έντονης κοινωνικο-οικονομικής κρίσης με την οποία έρχεται αντιμέτωπη η Ευρώπη. Υπάρχουν στη διάθεσή μας κοινοτικά οικονομικά μέσα τα οποία οι Ευρωπαίοι αλληλείς θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν όπως για παράδειγμα τα ήδη υπάρχοντα εργαλεία που προσφέρει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλείας ή προγράμματα εντός των προγραμμάτων πλαισίων έρευνας. Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω ακόμα μία φορά την κυρία Ιώτοβα για τη συνεργασία και για το γεγονός ότι συμπεριέλαβε στην έκθεσή της κάποιες από τις βασικές μου προτάσεις και ανησυχίες. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Τσουκαλά. Κύριε Τραμπαλή, θέλετε το λόγο. Κι εγώ να ευχαριστήσω την κυρία Ιώτοβα για τη συνεργασία και τη δυνατότητα να έχουμε ένα διάλογο για την προετοιμασία αυτής της εκθέσης. Ε, στην Επιτροπή εμείς εκφράσαμε στην τελευταία μάλλον συνάντηση τη θέση που έχουμε σε μια σειρά προτάσεων που γίνονται. Δεν χρειάζεται να πάμε παραπέρα από ό,τι έχουμε πει μέχρι τώρα και επίσης να ευχαριστήσω και τον κύριο Τσουκαλά για τις τροπολογίες που κατέθεσε οι οποίες σίγουρα ε, βελτιώνουν το κείμενο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ωραία. Με αυτό λοιπόν μπορούμε να περάσουμε πλέον στην ψηφοφορία. Ελπίζω να έχουν όλοι τις κάρτες τους. Καταρχάς ψηφίζουμε τη συμβιβαστική τροπολογία υπαριθμών 2. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. Εγκρίνεται ομόφωνα. πει υπολογία 8 και ψηφίζουμε την τροπολογία υπαριθμών 9 του κυρίου Τσουκαλά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. Εγκρίνεται ομόφωνα. Τροπολογία υπαριθμών 10. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση τη ψηφοφορίας. Εγκρίνεται ομόφωνα. Τροπολογία υπαριθμών 11 του κυρίου Τσουκαλά. Άρχεται η ψηφοφορία. πέρασε τη ψηφοφορίας. Εγκρίνεται ομόφωνα. Τροπολογία υπαριθμών 12 του κυρίου Τσουκαλά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία. Εγκρίνεται με 19 ψήφους υπέρ, 2 κατά. Καταπίπτει η τροπολογία υπαριθμών 13 του κυρίου Καντέκ και αρχίζει η ψηφοφορία για την τροπολογία υπαριθμών 14. Πέραση ψηφοφορίας εγκρίνεται. Άρχεται η ψηφοφορία για την 15. Πέραση ψηφοφορία. Εγκρίνεται ομόφωνα. Τροπολογία 16. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία. Εγκρίνεται ομόφωνα. Τροπολογία 17. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία. Συμβιβαστική τροπολογία υπαριθμών 3. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται ομόφωνα. Καταπίπτει 18. Ψηφίζουμε την 19. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. Εγκρίνεται και πάλι με μεγάλη πλειοψηφία. Τροπολογία 20. Άρχεται ψηφοφορία. Πέραση Πέρασε ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 4. Άρχεται ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία. Εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία. Καταπίπτουν 21 και 22. Ψηφίζουμε την τροπολογία 23. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 5. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία. πίπτη 24, ψηφίζουμε την τροπολογία 25. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία. Εγκρίνεται ομόφωνα. Ψηφίζουμε την τροπολογία 26, άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία. Ψηφίζουμε κατά τμήματα την τροπολογία 27. Πρώτο τμήμα, άρχεται η ψηφοφορία. Σε Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ένα σοσιαλιστή επιπλέον ψηφίζει. Ε? Εκτός μικροφώνου το σχόλιο. Συγγνώμη, δεν, είμαι, δεν ψηφίζω δυο φορές, αλλά έκανα λάθος ε, πατώντας το κουμπάκι. Τέλο πάντων, ούτω ή άλλω είναι μεγάλη διαφορά. Δεν θα αλλάξει τίποτα στη διαφορά. Είμαστε 13-8, οπότε εγκρίνεται. Στη συνέχεια, ε, έχει κάποιο αντίρρηση να ψηφίσουμε τις αιτιολογικές σκέψεις από την 1 ως 6 μαζί. Να τις ε, ψηφίσουμε από κοινού, λοιπόν. Διαφωνεί ο κύριος Ρωμαβαϊρόδα. Ε, εντάξει, εντάξει, αυτό σας ρώτησα. Τροπολογία 1, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ομόφωνα. Τροπολογία 2. Άρχεται ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία. Εγκρίνεται ομόφωνα. Τροπολογία 3. Άρχεται η ψηφοφορία. Σε σιέρα. Πέρασε ψηφοφορία. Ε, Εγκρίνεται. Τροπολογία 4. Πέραση ψηφοφορία. ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 6. Άρχεται η ψηφοφορία. Εγκρίνεται ομόφωνα. Συμβιβαστική τροπολογία 1. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας εγκρίνεται ομόφωνα, καταπίπτει 7 και ψηφίζουμε τώρα την έκθεση ως τροποποιήθηκε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. Εγκρίνεται ομόφωνα με 20 ψήφους, καμία αποχή. Συγχαρητήρια στην κυρία Ιώτοβα και σε όλους όσους συμμετείχαν στις συμβαστικές τροπολογίες. Να περάσουμε τώρα στο σημείο 5 της ημερήσιας διάταξης. Να σας πω απλώς ε, για το σημείο 4 ότι λογικά θα ψηφιστεί στην Ολομέλεια του Σεπτεμβρίου. Περνάμε στο σημείο 5 λοιπόν τη ημερήσια διάταξη. Αλλιευτικέ δυνατότητε και χρηματική αντιπαροχή που προβλέπονται στη Συμφωνία Αλλιευτική Σύμπραξη μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινου Ακροτηρίου. Ο Πάτε Κόμπ Γκάλαγκερ είναι εισηγητή. Παρουσιάστηκε ήδη η πρόταση και σήμερα ο εισηγητή θα μα παρουσιάσει το σχέδιο έκθεσή του. Να δώσω το λόγο λοιπόν στον εισηγητή για να μα ε, παρουσιάσει το σχέδιο έκθεση και κατόπιν θα λάβουν το λόγο και οι συνάδελφοι που θέλουν να συμμετάσχουν. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κάναμε μια σύντομη συζήτηση για το θέμα αυτό στην περασμένη συνάντησή μας. Πρόκειται για μια ε, ιδιαίτερη, αν θέλετε, ε, συμφωνία σε εταιρικής σχέσης. Πρόκειται για μια περιοχή υπερπεριφερειακή ε, εδώ Μαδέρα και όπως η Μαδέρα και η Κανάρη νήσι ε, και περιλαμβάνονται λοιπόν κάποιες ε, ειδικέ διατάξεις σχετικά τώρα όσον αφορά τα ε, Ηδη πρόκειται κυρίως για τόνο και κάποια πελαγικά και κάποια ε, βενθόβια ήδη αλλά όσον αφορά τις θέσεις εργασίας ε, πρόκειται για 10.000 περίπου θέσεις εργασίας και από εκεί και πέρα η σχετική ε, ε, εταιρεία η οποία διαχειρίζεται τα προϊόντα Υπάρχει μια αρχή, μια, ένας ε, θεσμός στο πράσινο κροτήριο που ασχολείται με τα θέματα αυτά. Καταλαμβάνουν ένα κάποιο μερίδιο, αν θέλετε, στι ε, στις ε, αγορές μετά της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου στέλνουν τα ψάρια. Αλλά εκτός από την Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν και σκάφη στην περιοχή από άλλες χώρες, παραδείγματος χάρη πω η Ιαπωνία, η οποία όμως δεν ψαρεύει παραδείγματος χάρη. Ε, είναι... Ε, εκεί ασχολείται με επισκευές σκαφών κτλ. Λόγω της ιδιαιτερότητας τώρα της συμφωνίας αυτής ε, υπάρχουν κάποιες δυσκολίες και κάποιες καθυστερήσεις υπήρξαν κενά αν θέλετε όσον αφορά τη, την στις συζητήσεις που γίνονται για τη συμφωνία αυτή το 2009 έγινε μια συζήτηση που εντόπισε πολλά προβλήματα και δυσκολίες που πρέπει να ξεπεραστούν. Από εκεί και πέρα υπάρχει ένα θέμα για... Ε, ε, υπάρχουν εκρεμή ζητήματα και όσον αφορά τα κτίρια ε, αποθήκευσης και όσον αφορά την υγειονομική κατάσταση αν θέλετε των κτίριων αυτών βεβαίως αποφελήθηκε η, το πράσινο ακροτήριο από τα κονδύλια που πήρε 385.000 βεβαίως υπάρχουν και τα τέλη για την αδειοδότηση και τα λοιπά ε, συνολικά Ανεβαίνει λοιπόν το ποσό 400 και κάτι χιλιάδες ευρώ και στο διάστημα 2007-2009 έχουμε καλύπτουμε αν θέλετε ε, με τα κονδύλια αυτά το 24% περίπου της, αναπτυ... της βοήθειας ή των κονδυλίων που παίρνει το πράσινο ε, ακροτήριο το νέο πρωτόκολλο έχουν αποφεληθεί λοιπόν οι πολίτες της χώρας αυτής το καινούριο πρωτόκολλο το οποίο ελπίζουμε να υπογραφεί θα βοηθήσει ε, περαιτέρω θα βοηθήσει τη βελτίωση των υποδομών για την παρακολούθηση τον έλεγχο των ενεργειών κτλ και θα επηρεάσει σημαντικά ίσως όχι σημαντικά αλλά θα επηρεάσει οπωσδήποτε και τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Η σύναψη λοιπόν του καινούριου πρωτοκόλου είναι πολύ σημαντική, θα καλύπτει ε, τις ζώνες στην δυτική ε, Αφρική και θα δώσει πέρα από αυτά που θα δώσει στο πράσινο ακροτήριο και ε, κάποια πλεονεκτήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται ε, για μια καινούρια διάσταση εδώ για κάποιες καινούριες περιοχές στη Δυτική Αφρική που μπορούν να χρησιμοποιήσουν και οι αλληλείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως εισηγητής θεωρώ ότι το καινούριο πρωτόκολλο είναι θετικό και για όλα τα συμβαλόμενα μέρη αν θέλετε και γι' αυτό συστήνω στην Επιτροπή να το εγκρίνουμε το πρωτόκολλο αυτό. Μιλάμε για πρωτόκολλο από την 1η Σεπτεμβρίου του 2011 έως το τέλος Αυγούστου του 2013. Ε, Καταρχήν, στην περασμένη μας συνάντηση συμφωνήσαμε κυρία Πρόεδρε ότι θα ψηφίσουμε για το θέμα αυτό τον Ιούλιο. Έκτοτε όμως όπως θα ξέρετε η Επιτροπή Περιβάλλοντος μας ζήτησε, συγγνώμη, η Επιτροπή Ανάπτυξης, όχι Περιβάλλοντος, μας ζήτησε να... Ε, αλλάξουμε το χρονοδιάγραμμά μας δεχτεί το δεχθήκαμε ε, όντως πήραν την τελευταία στιγμή τα σχετικά χρειάζεται λίγο παραπάνω χρόνο θα γνωμοδοτήσει η Επιτροπή Ανάπτυξης ε, όσον οπότε προτείνω να αναβάλουμε την ψήφιση από τον Ιούλιο το για το Σεπτέμβριο και αυτό δεν επηρεάζει τη συνέχεια της ειδική αυτής εταιρική σχέσης με, τον, με το πράσινο ακροτήριο. Δεν είναι τίποτα το τρομερό αυτό νομίζω όμως ότι είναι σημαντικό να ε, δώσουμε το χρόνο και στην, στις άλλες επιτροπές να γνωμοδοτήσουν και όμως πρέπει να βιαστούμε για να αρχίσει ήδη ω το δυνατόν πιο γρήγορα να ισχύει το πρωτόκολλο αυτό που είναι προς το συμφέρον και του Πρασίνου Ακροτηρίου και ε, προς το δικό μας συμφέρον. Και βεβαίως να μην ξεχνάμε και την συνιστόσα σχετίζεται με τα ανθρώπινα δικαιώματα εδώ και υπάρχει κάτι τέτοιο στο πρωτόκολλο. Ε, euh, Πρόεδρε, πολύ πολύ γρήγορα να συγχαρώ τον εισηγητή για τη δουλειά του και για την έκθεσή του. Σίγουρα οι ε, συμφωνίες αυτές για τον τόνο είναι πολύ σημαντικές για το κλάδο των Ξαλίας στην Ευρώπη η, συμφωνία αυτή είναι καλή, λειτουργεί καλά και είναι προς το συμφέρον της Ευρώπης αλλά σίγουρα και την ε, βοηθά και τη βιομηχανία μεταπής και τα λοιπά. Ε, θέλουμε λοιπόν ε, Πιστεύουμε ότι πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί ε, διατηρώντας βεβαίως τους αλευτικούς πόρους στην περιοχή και προ... θέλουμε να λειτουργεί και προς το συμφέρον του πράσινου ακροτηρίου. Για να μην σας καθυστερώ να πω ότι είναι μια καλή, πραγματικά καλή συμφωνία που αξίζει να την υποστηρίξουμε. Ο κύριος Καπούλα Ευχαριστώ. Εγώ ως ε, σκιώδης εισηγητής των σοσιαλιστών θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή για τα όσα μας παρουσίασε. Περιλαμβάνονται πάρα πολλές πληροφορίες, είναι εντελεχέστατα τα πάντα και ε, αναφέρονται πολύ σημαντικά θέματα. Θα ήθελα να πω εδώ ότι πρόκειται για μια Αφρικανική χώρα που είναι πολύ ιδιαίτερη. Υπάρχει δημοκρατία ε, με εναλλαγή στην εξουσία, δεν υπάρχει διαφθορά, γίνεται σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αυτή η Αφρικανική χώρα αποτερεί παράδειγμα καλής διακυβέρνησης. Ε, και πρόκειται λοιπόν για έναν από τους προτιμησιακού μα εταίρου. Στην έκθεση αναφέρονται τα βασικά ζητήματα, ε, ενισχύονται τα, ε, οι ενισχύσεις στον προπολογισμό προκειμένου να βελτιωθεί ο συγκεκριμένος τον νεμαίων στο πράσινο κροτήρι. Έχει συμπεριληφθεί και η πτυχή της βιωσιμότητας. Συμφωνούμε επίσης στο γεγονός ότι οι εργαζόμενοι επί των σκαφών θα πρέπει να είναι ε, από την ε, περιοχή και όχι απαρατήτως από όλη την περιοχή ΑΚΕ και Νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό ε, ενώπιον και των ε, ε, φαινομένων πειρατείας που έχουμε στις περιοχές. Υπάρχει μόνο ένα έλλειμμα εφαρμογής ε, ελέγχων και εποπτείας και πιστεύω ότι με τους επιπλέον αυτούς πόρους θα μπορέσουμε ίσως να πληρώσουμε και αυτό το κενό. Πρόκειται για καλή δουλειά. Ε, την οποία θα πρέπει να υποστηρίξουμε. Και θα ήθελα να ζητήσω από τους συναδέλφους μου να με συγχωρέσουν, αλλά επειδή πρέπει σύντομα να αναχωρήσω, ε, γιατί περιμένει το αεροπλάνο μου, θα ε, πρέπει να φύγω από τη συνεδρίαση. Δεν είναι έλλειψη σεβασμού, αλλά πραγματικά πρέπει να φύγω. Καλό σας ταξίδι, λέει η πρόεδρος, η κυρία Πατράο Νέβες. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Και εγώ με τη σειρά μου θα ήθελα να μιλήσω ως και όδηση για τη συγκεκριμένη έκθεση. Θα ήθελα καταρχάς να συγχαρώ το συνάδελφο Γκάλαγκερ για τα όσα έκανε. αντικατοπτρίζονται με πολύ ισορροπημένο τρόπο και οι θετικές αλλά και οι αρνητικές πτυχές και είχα ζητήσει το λόγο για να επισημάνω κάποιες πτυχές οι οποίες κατά την άποψή μου θα πρέπει ίσως να ε, τονιστούν λίγο περαιτέρω. Αναφερόμαστε σε μία μίεση των ετών. Από τα 4,5 χρόνια περάσαμε στα 3 χρόνια και ταυτόχρονα αυξήθηκε το οικονομικό αντιστάθμισμα. Αν κάνουμε το λογαριασμό έχουμε περάσει από, τα 270, από τις 270.000 ευρώ στις 330.000 ευρώ. Πρόκειται λοιπόν για μία ουσιαστική αύξηση, ε, κατά ένα τρίτο περίπου της 100 είναι η αύξηση και ε, έχει μειωθεί το χρονικό διάστημα στην οποία θα δοθούν τα κονδύλια. Θεωρώ ότι πρόκειται για ένα καλό στοιχείο, διότι ε, έτσι μπορούμε να υποστηρίξουμε τον αλλιευτικό τομέα στο πράσινο ακροτήρι και όπως ακούσαμε το πράσινο ακροτήρι αποτελεί καλό παράδειγμα χρηστής ε, πολιτικής διακυβέρνησης και η ανάπτυξή του ε, ήταν ε, πολύ σημαντική. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι χρειάζεται αυτή την υποστήριξη για να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε και ένα τομέα ο οποίος είναι και στρατηγική σημασίας για τη χώρα. Αυτό που έχει σημασία, όπως πάντα, είναι να υπάρχει όμως μιας κάποιος μορφής εποπτεία. Ένας κάποιος έλεγχος προκειμένου να μπορέσουμε να φροντίσουμε αυτό το οικονομικό ε, αντιστάθμισμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συνεισφέρει σε πραγματική ανάπτυξη του ελευτικού τομέα στο πράσινο ακροτήρι. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να αναφερθώ και σε κάποιες πτυχές ε, που περιλαμβάνονται στην έκθεση. Λέμε ότι το Κοινοβούλιο θα ζητήσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Μικτής Επιτροπής. Θα ζητήσει ετήσια αξιολόγηση και θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό το Κοινοβούλιο να μπορεί να παραστεί και στις συνεδριάσεις αυτές. Όλες αυτές οι πτυχές, καθώς επίσης και η ανάγκη να υπάρχει μια αιτήσια, ε, συγγνώμη, μια τελική αξιολόγηση για τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόστηκε το προηγούμενο πρωτόκολλο, είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη προκειμένου να συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την εφαρμογή του πρωτοκόλλου του Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το έχουμε πει επανειλημμένω, το Κοινοβούλιο έχει πλέον περισσότερες αρμοδιότητες και επομένω έχει σημασία να μπορεί και να ε, κάνει την κατάλληλη παρακολούθηση ένα επιπλέον στοιχείο τώρα. Εγώ θεωρώ ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να λαμβάνει πληροφορίε τακτικά για την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων. Υπάρχουν αρκετοί ε, πορτογαλικοί τομεί που ήρθαν σε επαφή μαζί μου διότι του ενδιαφέρουν ε, τα διάφορα πρωτόκολλα τα οποία συζητάμε εμεί εδώ με διάφορε χώρε. Το θέμα είναι ότι όταν φτάνουν σε εμά οι συμφωνίε ε, δεν γνωρίζουμε απαραίτητο τι συνέβη στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Είναι πλέον πολύ αργά και δεν ε, είναι πολύ εύκολο να ζητήσουμε οποιαδήποτε αλλαγή που θα μας επιτρέψει να αναθεωρήσουμε ίσως ε, μια συμφωνία και να φροντίσουμε και τα συμφέροντα των διαφορών κρατών μελών. Εάν όμως η παρακολούθηση ξεκινήσει εξ αρχής, θα μπορούμε να παρέμβουμε έγκαιρα με βάση φυσικά και τους όρους που προβλέπονται, προκειμένου να βελτιστοποιήσουμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό αυτές τις συμφωνίες και να είναι οι συμφωνίες προς όφελος ε, του Ευρωπαϊκού Αλληλευτικού Στόλου. Πρόκειται για σημαντικές πτυχές. Ε, Παρ' όλα αυτά θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Γκάλαχερ και να πω ότι αυτές οι πτυχές είναι σημαντικές και για αυτή τη συμφωνία αλλά και για τις μελλοντικέ συμφωνίες. Πρόεδρος, αυτό ακριβώς προσπαθούμε να κάνουμε και ξεκινήσαμε με τη συμφωνία με τη Μαυριτανία. Θα προσπαθήσουμε να ε, κάνουμε αντίστοιχα ε, πράγματα και με όλες τις ε, αλλιευτικές συμφωνίες. Πρόκειται για κάτι το οποίο ξεκίνησε και θα το συνεχίσουμε όπως έχουμε προβλέψει. Κύριε Λεβίν. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ και τον κύριο Γκάλαχερ για την έκθεσή του. Είναι σημαντικό και πολύ σωστό ότι τονίζετε στην έκθεσή σας πως ο έλεγχος και η παρακολούθηση μέχρι τώρα δεν λειτουργήσε πάρα πολύ καλά. Η ε, βάση της αξιολόγησης δεν λειτουργήσε καθόλου. Χαίρομαι λοιπόν που έγιναν κάποια πρώτα βήματα για να εφαρμοστεί ένα σύστημα ΕΜΕΣ στο πράσινο κροτήριο. Διότι πράγματι μέχρι τώρα δεν έγιναν μεγάλες προσπάθειες ε, να εξασφαλιστεί καλή εποπτεία και παρακολούθηση. Έγινε προσπάθεια να χρησιμοποιηθεί βέβαια η ακτοφυλακή, πράγμα το οποίο δεν απέδωσε καρπούς. Με άλλα λόγια δεν ε, υπάρχει ούτε έλεγχος αλλά δεν υπάρχει καν και αλλιευτική πολιτική στο πράσινο αυτό ακροτήριο. Οφείλουμε να πούμε γι' αυτό. Αυτό θα πρέπει να τονιστεί στο επόμενο πρωτόκολλο να τονιστεί ότι χρειάζεται ε, αλληλευτική πολιτική οποιαδήποτε πρόοδος επετεύθει επετεύθει λόγω των αρχών που ασχολούνται με την ανάπτυξη όχι λόγω μιας αλληλευτικής πολιτικής ε, επίσης όταν μιλάμε για τα αλληλευτικά αποθέματα και τα πλεονάσματα τα σχετικά. Είπε και ο, ο κύριος Κάλαχερ κάποια σχετικά. Υπάρχει υπάρχουν ανησυχίες εκεί για κάποια είδη μεταξύ των οποίων η θαλάσσια χελώνα παραδείγματο χάρη που, που απειλούνται από κάποια πράγματα που γίνονται πρέπει να τα δούμε λοιπόν και αυτά Επίσης, άκουσα αυτά που ελέγχουν για την α, ρήτρα διασφάλιση, για ρήτρα προστασίας των πόρων και για τα ε, ανθρώπινα δικαιώματα κτλ. Ωραία. Αλλά υπήρχαν προβλήματα με την κατάσταση που ισχύει σε κάποια σκάφη ε, και σε σχέση με τους εργαζόμενους και τα λοιπά. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε λοιπόν ότι και τα ευρωπαϊκά σκάφη που πάνε στην περιοχή πρέπει να συμμορφούνται με αυτές τις διατάξεις και σε όλα τα σκάφη που βρίσκονται εκεί. Ε, περιπτώσει η αυτές είναι όλες παρατηρήσεις που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας στην καινούργια συμφωνία. Το πλεόνασμα των, ε, πρέπει οπωσδήποτε να προσεχθεί ιδιαίτερα και θα πρέπει και η Ευρωπαϊκή Ένωση να φροντίσει να ελέγξει και να παραπάνω τις αρχές στο πράσινο ακροτήριο. Ευχαριστώ. Θα κάνω και εγώ την παρέμβασή μου. Δεν έχω να προσθέσω και πολλά. Όσον αφορά τους πόρους, θα ήθελα να πω ότι κυρίως είναι θέμα της ICAT, διότι το πράσινο ακροτήρι συμμετέχει στην ICAT και επομένω πρόκειται για ένα θέμα που δεν είναι τόσο πρόβλημα της συμφωνίας. Βέβαια δεν λέω ότι δεν έχει σχέση η συμφωνία γιατί όλα είναι αλληλένδετα, αλλά το θέμα αυτό είναι ε, πιο συγκεκριμένα θέμα της ICAT και να ε, τηρηθούν οι συστάσεις που έχει προτείνει η ICAT ε, για το θέμα αυτό. Από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η κυρία Μανουσοπούλου έχει το λόγο. <clears throat> Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πολύ σύντομα να πω με προσοχή διαβάσαμε την αξιολόγηση σημειώσαμε ό,τι έχει λεχθεί και είναι σαφές ότι όσον αφορά καταρχήν τη διοικητική λειτουργία αυτής της συμφωνίας ε, συναντήσεις της Μικτής Επιτροπής κυρίως, αλλά επίσης και τεχνικές συνεδριάσεις που χρειάζεται να γίνουν θα λάβουν χώρα πολύ πιο συστηματικά. Ε, το αποφασίσαμε αυτό, είναι στόχος μας για να ξεπεράσουμε αυτή το, την, ε, το χάσμα που υπήρχε στο διάλογο. Και εσείς θα λάβετε αμέσω κόπια ε, όποια έκθεση προκύψει από την Μικτή Επιτροπή. Τώρα, όσον αφορά τα άλλα ερωτήματα, για την συνέχεια που θα υπάρχει, ο έλεγχος που θα γίνεται, θα κάνουμε τα μέγιστα. Και σίγουρα η συμφωνία μπορεί να συμβάλλει με τα μέσα που έχει. Τα μέσα φυσικά από τη μια είναι πολύ λίγα. Ε, αυτές οι χιλιάδες ευρώ που έχουμε στη διάθεσή μας πραγματικά δεν είναι ποσά που θα λύσουν τα προβλήματα. Αλλά μπορούμε όμως να προσδιορίσουμε στόχους, να, δοθεί, ε, δοθούν συμβουλές, ε, να συμβάλλουμε. Και θα, ε, είναι πρόθεσή μας να το κάνουμε αυτό. Δεν θα είναι σίγουρα εύκολο, να επιβλέψει κανείς να, τη διαδικασία αυτή στο πράσινο ακροτήριο. Έχουμε κάποια μέσα και έχουμε τη θέληση να κάνουμε συγκεκριμένα μέτρα και να βελτιωθεί η κατάσταση. Επίσης, για τους παρατηρητές, το θέμα εδώ πέρα συστήνουμε στο πράσινο κρατήριο να υπάρχουν ε, άτομα που ελέγχουν στα απλία. Ε, Όλα αυτά είναι μέτρα τα οποία τα έχουμε στο μυαλό μας, είναι πρόθεσή μας, θα δώσουμε μια συνέχεια και φυσικά το θέμα των αποθεμάτων. Το είπε και η Πρόεδρος, αυτό θα εξαρτηθεί από αυτά, από την αξιολόγηση που θα μας δώσει το πράσινο κροτήριο. Αλλά φυσικά έχουμε την πρόθεση να δούμε να γίνουν κάποια βήματα και με, το δικό τους, ε, με δικά τους όργανα, με δικά τους ιστούτα, ούτως ώστε να βελτιωθεί οι, βελτιωθούν οι γνώσεις που έχουμε όσον αφορά τα αποθέματα. Αυτά σε γενικές γραμμές, αλλά σίγουρα έχουμε μπροστά μας πολλά να κάνουμε και σίγουρα δεν πετύχαμε ακόμα του, τους στόχους που θέσαμε. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Γκάλαγκερ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Καπούλα Σάντος, την κυρία Πατραονέβες ε, και τους άλλους συναδέλφους για τη συνεισφορά τους και να πω ότι όσον αφορά τις κοινέ συνεδριάσεις της Μικτής Επιτροπής, ε, το Κοινοβούλιο ενημερώθηκε και επιβεβαιώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, τώρα, αλλά αναφέρεται και στις παραγράφους 2 και 3 του σχεδίου έκθεσης, ε, το οποίο λέει ότι το Κοινοβούλιο θα ενημερώνεται πλήρως και αμέσως σε όλα τα στάδια της διαδικασίας που σχετίζονται με τη συμφωνία και την ανανέωσή του όπως ε, απαιτείται. Στη 2 και 3 παράγραφο αναφέρονται σαφέστατα αυτά. Βεβαίω θα θέλαμε να είμαστε σε θέση να παρακολουθούμε και να εποπτεύουμε πολύ πιο στενά, αλλά όπω μα είπε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είχαμε 60.000 ευρώ γι' αυτό, η αύξηση είναι πλέον στα 110.000 ευρώ και επομένω δεν θα γίνει και καμία πολύ μεγάλη αλλαγή. Βέβαια οδεύουμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Δεν είναι τέλειες βεβαίω όλες αυτές οι συμφωνίες, αλλά αυτό που θα πρέπει να διασφαλίσουμε είναι ότι κάθε φορά που ανανεώνεται κάποια συμφωνία ε, ή ακόμα και στη διάρκεια μια συμφωνία σε συνεδριάσεις που γίνονται επισημαίνουν ζητήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Πρέπει να είμαστε λίγο ρεαλιστέ και να ασχοληθούμε με τα θέματα αυτά, λαμβάνοντα υπόψη και το σύστημα υποπτία που διαθέτουμε. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει και μια αλληλευτική πολιτική συγκεκριμένη αλλά θα πρέπει να θυμάστε ότι δεν αφορά μόνο ευθύνε ε, των αρχών του Πράσινου Ακροτηρίου η συμφωνία αυτή. Είναι δυτή η διαδικασία και έχει και η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ευθύνε και ε, τα σκάφη που έχουν για να διασφαλίσουν άδειε θα πρέπει ναι, να είναι υπεύθυνοι, θα πρέπει να, να συνειδητοποιήσουν ότι το μέγιστο βιώσιμο απόθεμα είναι σημαντικό, αλλά αυτό θα πρέπει να το συνειδητοποιήσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι μόνο οι αρχές του πράσινου ακροτηρίου. Θα πρέπει λοιπόν να υποπτεύεται η κατάσταση όσο καλύτερα μπορεί, μπορούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σαφώς πρέπει να τηρηθούν και οι συστάσεις του ICAT και θα πρέπει όλα αυτά να εξετάζονται από κοινού. Πολλά από τα ζητήματα που ανέφεραν από όσους ε, παρενέβησαν θα συμπεριληφθούν στην έκθεση, τα έχω σημειώσει. Προτείνω λοιπόν το σχέδιο έκθεσης μαζί με τις τροπολογίες που μπορεί να προκύψουν στο ε, προθεσμία που θα δοθεί ε, για την κατάθεση τροπολογιών να εξεταστούν. Ναι, ευχαριστώ λέει Πρόεδρος. προθεσμία 20 Ιουνίου για την κατάθεση τροπολογιών το μεσημέρι στις 12 ψηφοφορία στην, Ευρωπαϊκή, στην Επιτροπή μας συγγνώμη. Θα γίνει βάσει των όσων είπε ο κύριος Γκάλακερ διότι δεν υπάρχουν κάποιες ενστάσεις. Θα περιμένουμε και τη γνωμοδότηση Επιτροπής Ανάπτυξης. Ελπίζω να έρθει κάποια στιγμή ε, η γνωμοδότηση. Ψηφοφορία 31 Αυγούστου στη συνεδρίαση που θα γίνει μετά από τις διακοπές του καλοκαιριού και στη δεύτερη ολομέλεια του Σεπτεμβρίου καταρχήν θα, πάει στην θα συζητηθεί το ζήτημα. Να ευχαριστήσω λοιπόν και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον εισηγητή. Ολοκληρώθηκε το συγκεκριμένο σημείο στην ημερήσια διάταξη και κατόπιν έχουμε το έκτο σημείο στην ημερήσια διάταξη, έκθεση του κυρίου Βαλέσα, γνωμοδότηση μάλλον, για την πράσινη βίβλο από τις προκλήσεις της ευκαιρίας προς ένα κοινό πλαίσιο στρατηγικής για τη χρηματοδότηση της έρευνας και της καινοτομίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή είναι η Επιτροπή Ήτρε. Η Επιτροπή Βιομηχανίας θέλει να εγκρίνει την έκθεσή της ε, στις 29 ε, Αυγούστου. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει το συντομότερο δυνατόν να διαβιβάσουμε και εμείς τη γνωμοδότησή μας. Τις ε, προάλλες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την πράσινη βίβλο και πλέον έχουμε τη συζήτηση της γνωμοδότησης. Να δώσω το λόγο στον κύριο Βαλέσα για να μας εξηγήσει τα της έκθεσής του, της γνωμοδότησής του, συγγνώμη, και στη συνέχεια θα δώσουμε το λόγο στους συναδέλφους και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος Βαλέσα έχει το λόγο. E, e, Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, το σχέδιο γνωμοδότησης που σας παρουσιάζω σήμερα σχετίζεται με την προσθήκη μια παραγράφου στο κείμενο της Επιτροπής Ήτρε μιας παραγράφου για συγκεκριμένη χρηματοδότηση της έρευνας και της καινοτομίας για την αλία ξέρουμε πολύ καλά ότι η αλία και η γεωργία είναι βασικοί πυλώνες της, ε, του ευρωπαϊκού οικοδομήματος χρειάζεται να τη στηρίξουμε ξέρουμε ότι στην Αλία υπάρχουν πολλά προβλήματα και η, η έρευνα είναι πραγματικά πολύ σημαντικό εργαλείο για να εξασφαλίσουμε στο μέλλον βιώσιμη αλία η πράσινη βίβλος εστιάζει την προσοχή της σε καινοτομία και νέες τεχνολογίες αλλά δεν περιλαμβάνει εδώ το χώρο της αλίας ήδη από την περασμένη φορά είχα πει ότι χρειάζεται άμεση ε, χρηματοδότηση για έρευνα στην αλία αλλά και στο, στο πρόγραμμα πλαίσιο, έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα δεν περιλαμβάνεται και εκεί τίποτε για, την, για έρευνα στη θάλασσα. Οπότε ε, θεωρούμε ότι υπάρχει κενό. Η, Ευρωπαϊκή Επιτροπή βεβαίως ξέρουμε ότι κάποιες προτάσεις μπορεί να κάνει αυτό το μήνα αλλά ε, πιστεύουμε ότι πρέπει να ενισχυθεί, να γίνει κάτι συγκεκριμένο για την έρευνα στον τομέα της αλίας και γι' αυτό προτείνουμε την προσθήκη αυτής της παραγράφου. Έχουμε στόχους στην αλία που δεν θα μπορέσουμε διαφορετικά να τους επιτύχουμε. Θέλουμε βιώσιμη αλία και σωστή βιομηχανική παραγωγή αλλιευτικών προϊόντων αν θέλετε. Δεν φαντάζομαι ότι χρειάζεται να σας παρουσιάσω επιχειρήματα για να σας πείσω. Τα ξέρετε όλοι αυτά. Γι' αυτό υποβάλλω το σχέδιο γνωμοδότησης και ελπίζω να το εγκρίνετε. Είναι μια προσθήκη λοιπόν στην έκθεση της ε, Επιτροπής Ήτρε. Χρειαζόμαστε συγκεκριμένα κονδύλια για συγκεκριμένους στόχους στον χώρο της Αλίας στην Ευρώπη. Ευχαριστούμε, κύριος Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, και να ευχαριστήσω και τον κύριο Βαλέσα για την ε, γνωμοδότησή του. Βιώνουμε θέματα λιτότητα. Πολλές χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή ε, έχουν οικονομικές πιέσεις και πολλές από τις αλληλευτικέ χώρες, όπως και η δική μου, κάνουν περικοπές στον προπολογισμό και φυσικά οι πρώτες περικοπές γίνονται στον προπολογισμό των επιστημών για την αλληλεία και ακριβώς αυτή τη χρονική συγκυρία, ακριβώ αυτή τη στιγμή η κυρία Δαμανάκη προτείνει να βελτιώσουμε την επιστήμη της αλίας. Αν θυμάστε καλά, οργανώθηκε και μία διάσκεψη που ε, περιελάμβανε τους ενδιαφερομένους και τους επιστήμονες και τους αλληλείς και προσπαθήσαμε να βελτιώσουμε τις σχέσεις μεταξύ των και να καταφέρουμε να συνεργαστούν καλύτερα. Είναι δύσκολο για μένα ως συντηρητικό από το Ηνωμένο Βασίλειο να ζητώ αύξηση του προϋπολογισμού. Ελπίζω να μην το πει κανένα στον επικεφαλής μου, αλλά εάν θέλουμε να βελτιώσουμε τα επιστημονικά δεδομένα και να έχουμε καλύτερα επιστημονικά στοιχεία, θα πρέπει να πληρώσουμε και το ανάλογο τίμημα. Ε, στη διάρκεια των συζητήσεων μας ε, για την ε, κοινή ελευθερική πολιτική, το είπαμε αυτό και θα πρέπει να ακούσουμε πολύ προσεκτικά αυτά που λέει ο κύριος Βαλέσα και να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη να χρηματοδοτήσουν την επιστημονική έρευνα για την αλία. Υπάρχει και το πακέτο μεταρρύθμισης ε, που αναφέρει συνεχώς η κυρία Δαμανάκη και το υποστηρίζω εγώ πλήρως. Θέλουμε να εξελιχθεί η διαχείριση και η ευθύνη στα κράτη-μέλη και στις περιφέρειες για τις περιφερειακές οργανώσεις αλίας και εγώ το υποστηρίζω πλήρως αυτό. Θεωρώ ότι θα πρέπει να καθοριστεί το πλαίσιο για να επιτευχθούν οι πλήρω οι στόχοι της κοινή αλληλευτικής ε, αλλά η καθημερινή διαχείριση θα πρέπει να είναι αρμοδιότητα των περιφερειών. Ήδη κάποιες περιφέρειες μας λένε πώς θα αντέξουμε το οικονομικό κόστος, θα υπάρξει επιπλέον κόστος για τον προπολογισμό και εμείς κάνουμε περικοπές στον προπολογισμό. Πώς λοιπόν θα αντέξουμε το κόστος αυτό. Και τώρα λέμε ότι θέλουμε να κάνουμε περικοπέ ε, στον προπολογισμό για την επιστημονική έρευνα. Αυτά τα δύο στοιχεία μπορεί να αποτελέσουν καταστροφή για το μέλλον της κοινή ελευθερικής πολιτικής και θα πρέπει να επιληθεί το πρόβλημα. Ο τρόπος να το κάνουμε είναι να ακούσουμε τα όσα έχει να μας πει ο κύριος Βαλέσσα. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Πατραονέβες. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Συμφωνώ πολύ με αυτά που είπε ο κύριος Βαλέσα και ο κύριος Στίβενσον. Φαίνεται ότι ακριβώς τη στιγμή που βρισκόμαστε ε, σε βαθιά νερά με την κρίση, ε, που υπάρχει επιπλέον ε, κόστος για τον προϋπολογισμό, αρχίζουμε να ζητάμε περισσότερα πράγματα για υποστημονική έρευνα και θα περικόψουμε τα στοιχεία, τον προπολογισμό λες και είναι κάτι το οποίο θα μας δώσει απευθείας αποτελέσματα. Αλήθεια είναι ότι δεν μας δίνει απευθείας αποτελέσματα, αλλά μας επιτρέπει να έχουμε βιώσιμη ανάπτυξη. Η αλληλεία, πολύ περισσότερο από άλλους τομείς, ε, εξαρτάται από τη βιώσιμη ανάπτυξη και αυτό φυσικά ε, πρέπει να βασίζεται και στην καλή επιστημονική έρευνα. Οποιαδήποτε περικοπή λοιπόν στο συγκεκριμένο τομέα θα μπορούσε να θέσει ένα αμφιβάλλο την ε, ε οικονομική σωστή οικονομική διαχείριση της αλληλείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον υπάρχει ένα επιχείρημα το οποίο ε, μόλις και οι συνάδελφοι και θα πρέπει να το δούμε λίγο πιο διεξοδικά. Γνωρίζουμε ότι η στρατηγική για το 2020 περιλαμβάνει μία σειρά από ιδέες για καλύτερη χρηματοδότηση και πιο πολλές δυνατότητες χρηματοδότησης. Και η αλία περιλαμβάνεται μεταξύ των στοιχείων της στρατηγικής για το 2020. Δεν θα πρέπει λοιπόν να χάσουμε αυτή τη χρυσή ευκαιρία που μας παρουσιάζεται αυτή τη στιγμή να προσπαθήσουμε να ζητήσουμε περισσότερα κονδύλια για την έρευνα για την αλία. Διότι αυτό ε, περιλαμβάνεται ε, στη στρατηγική το 2020. Ένα τελευταίο στοιχείο. Όλα αυτά φυσικά έχουν και κάποιο κόστος, το είπε πολύ σωστά ο κύριος Στίβενσον. Εάν θέλουμε λοιπόν να επενδύσουμε στην επιστημονική έρευνα, θα πρέπει να πληρώσουμε και τον οβολό μας, να αυξηθούν τα κονδύλια. Το θέμα είναι ότι η επιστημονική έρευνα θα αποδώσει καρπούς, αλλά όχι μεθοπρόθεσμα, ούτε βραχυπρόθεσμα, μακροπρόθεσμα. Έχει ναι μεν μία τιμή επιστημονική έρευνα, αλλά όλο αυτό το ποσό αποζημιώνεται διότι μας επιτρέπει να έχουμε βιώσιμη ανάπτυξη για τη διαχείριση της αλίας. Μεσοπρόθεσμα ή βραχυπρόθεσμα λοιπόν νομίζω ότι θα απολαύουμε τους καρπούς που μας ε, ε, υπόσχονται. Η κυρία Ιώτοβα. Πρόεδρε, Θα ήθελα να πω ως και εισηγήτρια ορισμένα πράγματα για το, η του κυρίου Βαλένσα. Θα ήθελα να τον ευχαριστήσω για τη θέση που παίρνει και ε, συμφωνώ με αυτό που λέει σε κάποια στιγμή ότι συγκεκριμένα χρήματα πρέπει να δίνονται για συγκεκριμένους σκοπούς. Είναι πράγματι αναγκαίων να ε, γίνεται κάτι τέτοιο και είναι σίγουρο ότι ε, αν θέλουμε να εξασφαλίσουμε ε, κάποια πράγματα για το μέλλον θα πρέπει να χρηματοδοτήσουμε να δώσουμε επιπλέον χρήματα για την έρευνα αν θέλουμε να ανταγωνιστούμε τους Ιαπωνέζους ή τέτοιες χώρες οι οποίες είναι πολύ πάρα πολύ πιο μπροστά από μας θα πρέπει να ενισχύσουμε τα κονδύλια με την, ε, που δίνουμε στην έρευνα. Θα πρέπει επίσης να προσέξουμε βεβαίως πώς γίνεται η διαχείριση αυτών των κονδυλίων. Δεν το αμφισβητώ. Αλλά και είδαμε ότι με τις νέες τεχνολογίες μπορούμε να εξασφαλίσουμε πολλά πράγματα όπως έχουμε πει σε παλιότερες εκθέσεις μας για όλους και για τους αλληλείς και για τους καταναλωτές και δεν μπορούμε να αγνοούμε το γεγονός ότι 70 εκατομμύρια περίπου άνθρωποι στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή ζουν, βρίσκονται στον τομέα της αλίας. Ευχαριστώ κυρία Λεβίν, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ και την, τον εισηγητή. Ε, πρόκειται για πολύ μεγάλο θέμα το στρατηγικό πλαίσιο για την χρηματοδότηση της έρευνας και της καινοτομίας. Δεν είμαι βέβαιη τι μπορούμε να χωρέσουμε σε όλο αυτό το καζάνι. Συμφωνώ πολύ με τις ε, παρατηρήσεις που αναφέρονται στη γνωμοδότηση. Αυτό που με κάνει να αναρωτιέμαι είναι κατά πόσον θα μπορούσαμε να κάνουμε πιο συγκεκριμένες προτάσεις. Ε, να δώσουμε κάποιες κατευθύνσεις ως προς τη μορφή της έρευνας που απαιτείται ε, όταν συζητάμε για παράδειγμα την διαχείριση της αλίας ή τη διατήρηση των υδάτινων αποθεμάτων. Νομίζω ότι δεν έχουμε και επαρκή στοιχεία σε θέματα συλλογής δεδομένων. Θεωρώ επίσης ότι δεν έχουμε και τα κατάλληλα μέσα για την ε, ε, εποπτεία και τον έλεγχο. Θεωρώ ότι έχουν γίνει καινοτομίες στο συγκεκριμένο τομέα που θα ήταν θετικέ για τον αλληλευτικό τομέα, αρκεί να μπορούσαμε να τις εφαρμόσουμε για να μπορέσουμε να πατάξουμε και την παράνομη λαθρέα και ε, άναρχη αλληλεία και να προαγάγουμε την νόμιμη αλληλεία που αυτό είναι που επιθυμούμε. Αυτό είναι αυτό το οποίο αναφέρεται σε οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο για το μέλλον της κοινή ελευτική πολιτικής και τη θαλάσσιας πολιτική, ότι χρειάζεται μια οικοσυμπριστομική προσέγγιση. Και εδώ δεν υπάρχει επιστημονική έρευνα. Πώς ε, επηρεάζεται ένα αλληλευτικό απόθεμα όταν έχετε το μέγιστη δυνατή απόδοση σε ένα άλλο, ε, αν υπάρχουν δυσκολίε, αν είναι ανελένδετα. όλα αυτά είναι ε, τμήματα ενός συγκεκριμένου θέματος το οποίο θεωρώ ότι χρειάζεται πολύ περισσότερη έρευνα για την αντιμετώπιση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και του αλευτικού τομέα εν γέννη μακροπρόθεσμα. Εάν λοιπόν μπορούσα μέσω τροπολογιών να κάνω κάποιες πιο συγκεκριμένες προτάσεις για το πού ακριβώς απαιτείται να γίνει έρευνα. Ε, θα μπορούσα να καταθέσω κάποιες τροπολογίες που θα γίνουν δεκτές. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να συγχαρώ τον συντάκτη της γνωμοδότησης, αλλά θα ήθελα να σταθώ και σε ένα ζήτημα που δεν ξέρω αν έχει συμπεριληφθεί επαρκώς στην έκθεσή σας. Αυτό είναι το θέμα της εφαρμοσμένης έρευνας. Καταρχά υπάρχει θέμα χρηματοδότηση. Όταν έχουμε περισσότερα χρήματα, σαφώ θα μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε περισσότερα προγράμματα. Παλιά θεωρούσαμε ότι όταν η χρηματοδότηση της, ε, ε, του ελευτικού τομέα ήταν στον προπολογισμό για την αλληλεία, ήταν πολύ καλύτερα προσαρμοσμένη από τώρα που βρίσκεται στον προπολογισμό για την εφαρμοσμένη έρευνα. Από τότε που βρίσκεται στο πρόγραμμα πλαίσιο διαπιστώνουμε ότι αυτό που πρημοδοτείται είναι η έρευνα αριστείας και όχι η εφαρμοσμένη έρευνα και τελικώς το μεγαλύτερο τμήμα της απαραίτητης χρηματοδότησης για την αξιολόγηση των πόρων και ούτω καθεξής δεν περιλαμβάνεται στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο γιατί πρημοδοτείται η έρευνα αριστείας. Ε, το είπαμε 20 φορές σήμερα. Αυτή είναι και η έρευνα που μας ενδιαφέρει λιγότερο στον τομέα της αλληλείας και γι' αυτό ακριβώς ε, ε, πλήττονται και οι ερευνητές ε, των αλλιευτικών Ινστιτούτων. Δηλαδή, εάν δεν δημοσιεύσουν ε, τα δεν ξέρω ποια πράγματα για τα γνωσμένου κύρους περιοδικά, πέφτουν σε δυσμένεια ακόμα και στη χώρα τους, διότι δεν κάνουν την κατάλληλη έρευνα. Αυτό το οποίο λοιπόν θα ήθελα να επισημάνουμε και αυτό νομίζω ότι αναφέρεται και στην έκθεση του εισηγητή της Επιτροπής ΙΤΡΕ, της εισηγήτριας, συγγνώμη, είναι τι είδου έρευνα χρειάζεται για την ε, κάθε πολιτική. Και σε αυτή την περίπτωση μιλάμε για την αλληλευτική πολιτική. Επιμένω ότι δεν μας ενδιαφέρει η έρευνα αριστείας που ε, τονίζεται τόσο πολύ στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο, αλλά η εφαρμοσμένη έρευνα που δεν χρησιμοποιείται τόσο πολύ στην παρούσα έρευνα και στη χρηματοδότηση τη έρευνα ε, στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο θεωρώ ότι είναι ένα στοιχείο το οποίο θα πρέπει να λάβουμε υπόψη. Επιπλέον των όσων είπε και η κυρία Λεβίν, με την οποία συμφωνώ απολύτω. Η έρευνα αυτή τη στιγμή επικεντρώνεται στα οικοσυστήματα και αυτή είναι μια έρευνα η οποία είναι εκ διαμέτρου εντίθετη, είναι πολυτομιακή και απαιτείται μια προετοιμασία και κάποιε γνώσει που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν και έτσι δεν υπάρχουν αποτελέσματα. Πράγματι λοιπόν είναι ένα πολλά προβλήματα τα οποία επαναλαμβάνουμε συνεχώ και τελικώ αυτή η έρευνα δεν μα βοηθά σε καμία περίπτωση. Πρόκειται λοιπόν για ένα από τα θέματα τα οποία θα πρέπει να λάβουμε υπόψη αν θέλουμε η οικοσυστημική προσέγγιση να ε, είναι βιώσιμη και να μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη. Να δώσουμε τώρα το λόγο στον κύριο Φούξ από τη Γενική Διεύθυνση Έρευνας. Good afternoon. Καλησπέρα σας. Αντικαθιστώ τον συνάδελφο ο οποίος δεν μπόρεσε δυστυχώς να έρθει σήμερα, αλλά και εγώ ασχολούμαι με την ε, έρευνα και με τη χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων του 7ου προγράμματος πλαίσιου θα, όπως σας είπαμε και την περασμένη φορά βεβαίως είναι πολύ νωρίς τώρα να πάρουμε οποιασδήποτε αποφάση για τη χρηματοδότηση για το επόμενο στρατηγικό πλαίσιο. Συζητήσεις έχουν αρχίσει αλλά αποφάσεις δεν έχουν πάρθει και επειδή θα Βεβαίω τις συζητήσεις θα προσέξουμε και ιδιαίτερα αυτά που λέγονται στην πράσινη βίβλο. Ε, η αλληλεία περιλαμβάνεται στο κομμάτι για την ασφάλεια των τροφίμων και την περασμένη ε, Παρασκευή είδαμε ε, που, ε, ότι ενδιαφέρεται ή, υπήρξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για μια συνδιάσκεψη που έγινε σχετικά με τη μελλοντική έρευνά μας και χαιρόμαστε γι' αυτό επίσης Σημειώσαμε αυτό που είπατε για πολλά από αυτά που είπατε. Βεβαίως χρειάζεται η έρευνα στην αλλή, αλλά σημειώστε ότι δεν ξεκινούμε από το μηδέν έχει ήδη έχουν γίνει ήδη με τεράστιες προσπάθειες και ήδη στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο συνολικά 25 εκατομμύρια ευρώ διατίθεται ε, για τον τομέα τον οποίο συζητάτε αυτή τη στιγμή. Ο, ο, Βεβαίω δεν χρηματοδοτούμε μοναχά βασική έρευνα, θεωρητική έρευνα, αλλά καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να ε, βοηθήσουμε τον κλάδο πιο πρακτικά. Και γι' αυτό ζητήσαμε ε, να υπάρχουν και κονδύλια για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πιστεύουμε ότι αυτό θα βοηθήσει Επίσης πιστεύουμε ότι χρειάζεται μεγαλύτερος συντονισμός μεταξύ των κρατών μελών στα, στην έρευνα. Ε, αναφέρθηκε η οικονομική κρίση την οποία βιώνουν τα περισσότερα κράτη-μέλη. Αν θέλουμε λοιπόν να είμαστε στην έρευνα πιο αποτελεσματικοί θα πρέπει να αποφύγουμε επικαλύψεις και να υπάρχει καλύτερος συντονισμός. Και τελικά για την εφαρμοσμένη έρευνα που είπατε κυρία Πρόεδρε είναι ενδιαφέρουσα η συζήτηση αυτή θα μπορούσαμε να την κάνουμε κάποια στιγμή αλλά ήδη προσπαθούμε να βρούμε μια κάποια συνέργεια και συμπληρωματικότητα μεταξύ του ε, του 7ου προγράμματος πλαισίου και του νέου ταμείου αλίας το οποίο δημιουργείται γιατί πιστεύουμε ότι οι δύο αυτοί οι θεσμοί, αν θέλετε, οι δύο αυτές προσεγγίσεις είναι συμπληρωματικές και κλείνοντας θα ήθελα να σας συγχαρώ για όλη τη δουλειά που έγινε στο θέμα αυτό και να σας ευχαριστήσω για τη στήριξή σας στην έρευνα. Θέλετε να προσθέσετε κάτι κύριε Βαλέσα. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συμμετείχαν στη σημερινή συζήτηση. Θα ήθελα να ζητήσω από όλους να καταθέσουν τροπολογίες για την ε, γνωμοδότησή μου. Να σας υπενθυμίσω βεβαίω ότι αυτή η πράσινη βίβλος είναι πολύ περίπλοκη. Δεν ξέρω τι θα μπορέσουμε να κάνουμε και τι θα μπορούσαμε να συμπεριλάβουμε ε, εμείς ως Επιτροπή Αλία στην έκθεση της Επιτροπής ε, Βιομηχανίας. Εμείς θα πρέπει να φροντίσουμε να υπάρχει καλύτερη μεταχείριση για την αλληλεία από τη μεταχείριση που έχει στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο και να φροντίσουμε να μην μας κλείσουν την πόρτα στη κατάφατσα όπως μας έκαναν και στο παρελθόν. Θα ήθελα λοιπόν να αναφέρετε μία φράση τουλάχιστον στην έκθεση αυτή, η χρηματοδότηση των επενδύ... της έρευνας για την αλία. Αυτό λοιπόν και σας καλώ να καταθέσετε τροπολογίες. Ευχαριστώ πολύ. Να πω μόνο ότι η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών είναι 20 Ιουνίου στις 12 το μεσημέρι και ψηφοφορία στην Επιτροπή Αλίας θα έχουμε στις 12 Ιουλίου και στην Επιτροπή Ήτρε ε, στα τέλη του Αυγούστου. Δεδομένου ότι πρόκειται για γνωμοδότηση και πρόκειται για ένα θέμα το οποίο μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα, θεωρώ ότι όλοι εδώ θα ε, θέλαμε να ληφθεί υπόψη δεόντω το ζήτημα. Αυτό που θα πρέπει να δούμε με τον κύριο Βαλέσα είναι πώ θα μπορέσουμε οι θέσει που θα εγκρίνουμε εμεί εδώ να περάσουν υπό τη μορφή τροπολογιών ε, στην έκθεση της εισηγήτριας ε, στην Επιτροπή Βιομηχανίας. Έτσι ίσως θα μπορέσουμε να περάσουμε το μήνυμά μας. Θα δούμε πώς θα γίνει το ζήτημα, διότι οι γνωμοδοτήσεις χωρίς λόγο είναι άχρηστες, είναι κενό γράμμα. Ε, μισό λεπτό θα ολοκληρώσω, θα σας δώσω το λόγο. Το να έχουμε μία έκθεση με μία σειρά από τροπολογίες λοιπόν που θα εγκριθεί ε, είναι ίσως η πιο κατάλληλη λύση. Μπορεί να είναι τροπολογίες δικές σας εξ ονόματος Επιτροπής Αλίας ε, στην ε, γνωμοδότηση της κυρίας Μαρίσα Αματίας στην Επιτροπή Ήτρε. Σας δίνω το λόγο. Εγώ έπρεπε να κάνω το σχόλιο μου αλλά τέλος πάντων να σας δώσω το λόγο. Ξέχασα να σας πω ότι είχα μια πολύ επικοδομητική συνάντηση με την κυρία Ματίας και είναι ανοιχτή στις προτάσεις μας. Νομίζω ότι μπορούμε λοιπόν να θεωρήσουμε ότι θα μπορέσουμε ίσως να περάσουμε τις τροπολογίες μας. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Το θέμα είναι να βρούμε ποια είναι η κατάλληλη διαδικασία προκειμένου να συμπεριληφθούν οι τροπολογίε αυτέ στο κείμενο τη κυρία Ματίας. Με αυτό λοιπόν ολοκληρώνεται και το έκτο σημείο στην ημερήσια διάταξη και στη συνέχεια έχουμε το σημείο υπαριθμών 7 το οποίο είναι και κλεισμένο των θυρών και έχουμε συζήτηση για την εξωτερική πολιτική με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήθελα να ζητήσω από όσου όσους δεν επιτρέπεται να βρίσκονται στην αίθουσα να βγουν